en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion. μελλοντική προεδρία και εν ώψη τη μελλοντική μάλλον προέδρου θα προσπαθήσω να μιλήσω στα γαλλικά. Σας προειδοποιώ. Ό,τι λέτε αυτή τη στιγμή αναμεταδίδεται άμεσα στο διαδίκτυο. Εγώ είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος της παλιάς ε, επιτροπής, αλλά δεν θα έχω το ίδιο αξίωμα στην θητεία αυτή. Εγώ απλώς έχω τον ρόλο να εγκαθιστήσω στο θόκο του Προέδρου, τον μέλο τα πρόεδρο ή την πρόεδρο, δεν ξέρω, θα δούμε. Έχουμε απαρτία, δείχνει μάλλον. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει μια υποψηφιότητα για πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, παρακαλώ. Η κυρία Κρέζα. Les boutons, c'est le plus important, n'est-ce pas? Ah, donc, euh, Αν βρω το σωστό κουμπί, ε, λέγομαι Κατρίν Κρέσ από την ομάδα του Προσένου, εξωτερών της ομάδας μας, θα ήθελα να την υποψηφιότητα μιας υποψηφίου, της κυρίας Εύα Ζουλή. Et la candidate Πρόεδρος, συμφωνεί η εν λόγω ε, υποψήφιος. Μάλιστα, δέχομαι την υποψηφιότητα με μεγάλη χαρά, πρόεδρε. Α, με χαρά. Ωραία, και εμείς, και εμείς χαιρόμαστε. Τώρα φαντάζομαι θα έχετε ε, συμπληρώσει το έγγραφο που αφορά τα οικονομικά σας συμφέροντα. Πατάτε και το κουμπί για να σας ακούω. Μάλιστα, μάλιστα, το συμπλήρωσα, συμπλήρωσα αυτή τη δήλωση. Τα, της μετοχής σας στην Έλφα Τικητέν. Όχι, πρόεδρε, δεν έχω πια εδώ και πολύ καιρό εκεί μετοχές. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Άλλες υποψηφιότητες. Διαδικαστικό. Ο κύριος Μαρτινές. Quand je suis εγώ όταν προσπάθησα να πάρω το σωστό, το σωστό κανάλι εδώ, άκουγα δεν να ακούω ισπανικά, ακούω γερμανικά. Δεν ξέρω. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να πούμε στον τεχνικό. Γιατί έχουμε ταυτόχρονα δύο φωνές. Το πρόεδρο και ταυτόχρονα την γερμανική διερμηνία. Στο κανάλι μηδέν, Δεν ξέρω αν ο μόνος είμαι. Α μην μα απασχολεί αυτό, λέει ο πρόεδρο τώρα. Μια που υπάρχει μόνο μία υποψήφιο, εάν καθένα δεν θέλει μυστική ψηφοφορία, που δεν νομίζω ότι θέλει κανένα, μπορούμε να σας πω κύριε Ζολή ότι θα έχετε μια περίοδο ως πρόεδρο Και... Ε, τώρα, τώρα. Ζούμε, λέω, μια δύσκολη περίοδο για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών επιθέσεων. Οικονομική κρίση, κλιματολογική κρίση. Δεν είχαμε ποτέ μια τόσο δύσκολη περίοδο για να πετύχουμε του στόχους της χιλιετίας. Θα το κάνετε μαζί μας εδώ. Και εδώ είμαστε μεταξύ μας όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε υπέρ ενός ισχυρού ρόλου της Ευρώπης για την ανάπτυξη και για η κοινωνική δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Θα το κάνετε αυτό. Εσείς ε, γράψατε ένα βιβλίο που λέγεται «Δικαιοσύνη υπό ε, Development under siege, ε, dernière page sera heureuse υποκατάληψη. Ε, διαβοής νομίζω ψηφοφορία. Οπότε θα μπορέσω να παραδώσω το θόκο αυτό με μεγάλη φορήση σε κάποιον άλλον. Με μεγάλη συγκίνηση δέχομαι αυτή την θέση. Ξέρω ότι σε όλο το κοινοβούλιο δεν υπάρχει πιο σημαντική επιτροπή από αυτή εδώ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αντιμετωπίζουμε πολλαπλά προβλήματα των κλιματολογικών αλλαγών και των θυμάτων που υπάρχουν γι' αυτό στις άλλες χώρες. εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Χιλιάδες δισεκατομμύρια θα χρειαστούν και δεν έχουμε αυτούς τους πόρους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, το σύνολο της αναπτυσιακής βοήθειας στον κόσμο είναι 100 δισεκατομμύρια περίπου και αυτό είναι τελείως ανεπαρκές για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές των κλιματολογικών αλλαγών. Ο κίνδυνος είναι να θυσιαστεί η ανάπτυξη για το κλίμα και να θυσιαστεί η ανάπτυξη για την οικονομική κρίση. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η οικονομική κρίση θα εμβαθυνθεί ακόμα, θα επιδεινωθεί, θα διαρκέσει. Και εργασία μας είναι να ευιστοποιήσουμε τους ε, συμπολίτε μας στο γεγονός ότι η ανάπτυξη έχει προτεραιότητα. Αυτό είναι το έργο που θα πρέπει να επιτελέσουμε τα πέντε επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να παρουσιάσω αυτόν λιγάκι πριν εκλεγώ ευρωβουλευτής τα τελευταία 7 χρόνια ήμουνα στην υπηρεσία της ε, ε, νορβηγικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη, ιδίως για τη δημιουργία ενός ε, οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης, τους φορολογικούς παραδείσους και το πλήσιμα βρώμικου χρήματος. Πριν ήμουνα 20 χρόνια στην, στην τοπική διοίκηση στη Γαλλία Ελπίζω, ελπίζω ότι η πείρα μου θα βοηθήσει για να μπορέσουμε καλά να εργαστούμε αυτά τα επόμενα πέντε χρόνια. Τώρα θα περάσουμε στην εκλογή των τεσσάρων αντιπροεδρών της Επιτροπής αυτής. Λοιπόν, έλαβα μία υποψηφιότητα, τις εξής υποψηφιότητες μάλλον, για τους αντιπρόεδρους. Πρώτος Πρώτη αντιπρόεδρος, η κυρία Στίφλερ. Είναι παρούσα η κυρία Στίφλερ. Δεχόσαστε να γίνετε πρώτη αντιπρόεδρος. Μάλιστα, δέχομαι την πρόταση αυτή αυτή την εντολή και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να δεχθώ στο ύψος των περιστάσεων. Πρόεδρος, συμπληρώσατε τη δήλωση για τα οικονομικά σας φέροντα, μάλιστα. Πρόεδρος, άλλη υποψήφοι ως πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Όχι. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε την κυρία Στίφλερ διαβοής. Κυρία Στυφλέρ, μπορεί να έρθει να κάτσει εδώ δίπλα μου. Έλαβα την πρόταση της υποψηφιότητας του κυρίου Ντέβα ως δευτέρον του Προέδρου. Ο κύριος Ντέβα είναι παρόν. Δεχόσαστε την υποψηφιότητα αυτή ως δευτέρον του Προέδρου της Επιτροπής μας. Μάλιστα, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα αναλάβω το αξίωμα αυτό. Πρόεδρο, συμπληρώσατε την δήλωση των οικονομικών σας φερόντων. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρο, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για τη θέση αυτή. Εάν όχι, προτείνω να εκλέξουμε τον κύριο Ντέβα ως δεύτερον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης διαβοής. Καλό τον κύριο Ντέβα να κάτσει εδώ μπροστά στο Προεδρείο. Thank you. J'ai reçu la proposition de la nomination de... Κατόπιν έχουμε την πρόταση της υποψηφιότητας του κ. Σενική ως τρίτου αντιπρόεδρου της Επιτροπής μας. Α, συγγνώμη, η κυρία, η κυρία. Η κυρία είναι παρούσα? Μάλιστα, εδώ είμαι. Δεχόσαστε την υποψηφιότητα αυτή, τρίτη αντιπρόεδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, δέχομαι. Α, καλά είναι να χρησιμοποιώ και το μικρόφωνο. Ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, να μπορώ να συμμετάσχω στην επιτροπή αυτή τόσο δύσκολη. Θα καταβάλω για κάθε προσπάθεια. Στο μου θα μου δώσετε. Ευχαριστώ. Λέει Πρώτα, διπληρώσατε τη δήλωση των οικονομικών σας συμφερόντων. Μάλιστα. Ωραία. Άλλε υποψηφιότητες για την θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Αν όχι, να περάσουμε στην ε, εκλογή τη κυρία Ανίκη με ε, βοή, Και καλό την κυρία Ζανίκη να έρθει να κάτσει εδώ δίπλα μας στο Προεδρείο. Έλαβα μια πρόταση υποψηφιότητα της κυρία Κρετού ω τετάρτη αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης. Η κυρία Κρετού απουσιάζει αλλά μας έγραψε μια επιστολή, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Μαρτινές μπορεί να μας διαβάσει, μπορεί να μας ενημερώσει. Όχι, δεν θα σας διαβάσω την επιστολή, απλώς θα να σας πω ότι η κυρία Χρυσού δεν μπορούσε να είναι παρούσα για πολύ σημαντικούς εικονιακούς προσωπικούς λόγους και μας ζήτησε μια που είναι υποψήφιση της ομάδας να υποβάλουμε την υποψηφιότητά της στην τελευταία θητεία ήταν ενεργό μέλος της Επιτροπής αυτής και δέχεται ευχαρίστως, είναι ενθουσιώδης για την υποψιότητα για την Προεδρία αυτή, ε, συμπλήρωσε την ε, σχετική δήλωση για τα οικονομικά της συμφέροντα. Και με χαρά κάνω αυτή την παρουσίαση έξω των ξενομετρήσεις. Η επιστολή έχει αποστέλει σε εσά ω πρόεδρο τη Επιτροπή. Ναι, μάλιστα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε δέχεται λοιπόν αυτή την υποψηφιότητα, τετάρτη σαν πρόεδρο. Γραπτό, με επιστολή. Ναι, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε για τη θέση αυτή η τετάρτη του αντιπρόεδρου. Όχι. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στην εκλογή της κυρίας Κρυσίου διαβοής. Λοιπόν, τελειώσαμε την συγκρότηση σώμα της Επιτροπής μας με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρος και προτείνω μια που θα συνεργαστούμε καταρχήν δυόμιση χρόνια και μετά άλλα μισή χρόνια να παρουσιαστούμε οι μεν στους δε. Μπορούμε ο καθένας ένα λεπτό να πάρει για να πει ποιος είναι, από πού προέρχεται και ποιες είναι οι ελπίδες και τα οράματά μας. Euh, euh, θα les ranger comme ça et on peut commencer euh, par... Euh, Μπορούμε να αρχίσουμε με τα έδρανα, να αρχίσουμε από εσά. Ένα λεπτό καθένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μωρή Πόγκα. Έχω ε, εκλεγεί στα ευρωπαϊκά διαμερίσματα από τον Ειρηνικό και είμαι και ειρηνικό άνθρωπο. Πριν ήμουν υπεύθυνο ε, ως μέλος κυβέρνησής μου επί 10 χρόνια. Τώρα προήχθη εις Ευρωβουλευτή. Τι περιμένω από την Επιτροπή μας. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να κοιτάξει ιδιαίτερα το θέμα της ε, σύνδεσης, του καθεστώς σύνδεσης σχέσεις δηλαδή της Ένωσης με τις μικρές χώρες του ειρηνικού, τα υπερπόντια διαμερίσματα κλπ. Γιατί ορισμένες χώρες μέγκη της Ένωσης έχουν τέτοια τμήματα όπως η Γαλλία. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το καθεστώς αυτών των περιοχών, ΠΤΕΜ όπως λένε στα γαλλικά. Ευχαριστώ. Μπορείτε να είστε καθιστή όταν θα αυτό παρουσιαζόσετε, γιατί βοηθάει αυτό και για την, ε, τις κάμερες και για τον ήχο. Έκανε ένα λάθος, ε, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε του αντιπρόεδρους, γι' αυτό παρακαλώ να συνεχίσουμε του αντιπρόεδρους και μετά επανερχόμαστε στην αίθουσα. Πρώτη αντιπρόεδρος, θα είμαι σύντομη. Λέγομαι Μισελ Στίφλερ, είμαι αντιδήμαρχο τη Μιλού στην Λασατία. Είμαι μέλο τη σύγχρονης αριστεράς υπό λοιπόν, το Ζαμαρί Μποκέλ. Είμαι βουλευτής εδώ και μερικές μέρες, ευρωβουλευτής εννοώ. Έχω σπουδάσει φαρμακοποιός. Δεν είναι πολιτικό βέβαια αυτό, αλλά τελικά δεν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά και θα δώσω το λόγο στο γείτονά μου, εκτός αν κάποιος χρειάζεται επιπλέον πληροφορίε αν θέλετε ρωτήστε με. Λέγουμε Nerds Diva. Συνεδριάζω στην Επιτροπή αυτή εδώ και 10 χρόνια. Δύο κοινοβουλευτικέ θητείες. Είναι σημαντική επιτροπή. Ήμουν συντονιστή τη ομάδα ΕΛΚ Ευρωπαίοι Δημοκράτε, με μία συνάδελφο τα τελευταία πέντε χρόνια στην Επιτροπή ανάπτυξη και την ε, Επιτροπή Αντιπροσωπεία ΑΚΕ. Δεν είμαι στην ομάδα αυτή πια για λόγους που δεν τους ελέγχω εγώ. Είμαι μέλος μιας νέας ομάδας, συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, συντονιστής. Πριν έρθω στο Ευρωκοινοβούλιο μου είμαι ένα μέλος του, της Βρετανικής Βουλής και της Βρετανικής Κυβέρνησης υπό τον Τζον Major. Έχουμε μεγάλες, τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας, όπως είπε και η Πρόεδρος και ο προηγούμενος Πρόεδρος. Μεγάλες προκλήσεις σε όλο τον κόσμο και ως προς την ανάπτυξη και ζούμε και την οικονομική κρίση και πρέπει να δώσουμε μεγάλες μάχες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πιο φτωχούς στον κόσμο. Μεγάλη πολιτική μάχη αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζανίκη, λέγομαι Ήβα Τζανίκη, είμαι Ιταλίδα. Δεν έχουμε μεγάλη πολιτική ζωή γιατί προέρχομαι από τον κόσμο του θάματο, που δούλεψα 45 χρόνια, τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Συνάντησα ένα σωρό κόσμο, σημαντικού ανθρώπου. Πήρα πάρα πολλά από τη ζωή και κάποια στιγμή είπα, ε, ήρθε η στιγμή να δώσω κι εγώ κάτι. Δεν ξέρω αν διάλεξα το σωστό δρόμο. Σίγουρα στη σωστή επιτροπή τη διάλεξα. Με πάθος, με αγάπη, όπως πάντα έκανα, θα φροντίσω να δράσω και εδώ υπό την καθοδήγηση της Προέδρου μας, των άλλων εμπειρών συναδέλφων. Συνήθως ο κόσμος που προέρχεται από τον κόσμο του θάματος αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και το καταλαβαίνω αυτό, αλλά επειδή η οικία μου είναι αυτή που είναι, όπως τη βλέπετε, είναι εγγύηση. Δεν είμαι κοπελίτσα. Θα δώσω ό,τι μπορώ. Σας ευχαριστώ όλους για το πνεύμα συνεργασίας και εύχομαι καλή δουλειά και καλή συνεργασία γιατί τη χρειάζομαι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ξαναγυρίζουμε στην αίθουσα. Παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας γιατί είμαστε πολλοί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν σας χαίρομαι για την εκλογή σας και τους αντιπρόεδρους. Λέγομαι Γκέι Μίτσελ, με μέλος του ΕΛΚ, από κοινού συντονιστή με τον κύριο Κάσμαρα. Ήμουν μέλος της ίδιας επιτροπής του προηγούμενου κοινωνίου, συγγετής για το ε, εργαλείο ανάπτυξης και συνεργασίας που είναι ο βασικός νόμος, ας το πούμε, για την ανάπτυξη βοήθεια. Είπε επίση και τον ε, επίγουση επιστημιστική βοήθεια εισηγητή, ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ήμουν πρώην Ιρλανδός βουλευτής και υπουργό εξωτερικών κάποια στιγμή στην κυβέρνηση της Ιρλανδίας. 11 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια πεινάνε και υπάρχουν ένα σωρό άλλα εκατομμύρια κόσμος που δεν έχουν καθαρό νερό. Ελπίζω όλοι να συνεργαστούμε, να, να φροντίσουμε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Είμαι. Ολονός ευρωβουλευτής. Τα τελευταία πέντε χρόνια σε αυτή την επιτροπή. Θεωρώ αυτή την επιτροπή πολύ σημαντική. Τα τελευταία πέντε χρόνια κυρίως κατέβαλα προσπάθειες ώστε οι χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλέκονται εντονότερα στην αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν κάνω λόγο για τις καινούργιε χώρες, αλλά για εκείνες τις χώρες που δεν είναι και επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέλη σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να ληφθεί αυτό υπόψη. Ήμουν και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στις τοπικές άρχες και κοινότητες εκπρόσωπος. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. My name is Σα ευχαριστώ. Είμαι Ούγγρο Ευρωβουλευτή, νέο μέλο σε αυτή την ε, επιτροπή, αλλά όχι καινούριο Ευρωβουλευτή. Ήμουν στην παλαιά θητεία και προηγούμενα ήμουν και μέλος ε, ε, στην, Βουλή της Ουγγαρίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ξέρω ότι είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή και θέλω να είμαι χρήσιμο ως μέλος σε αυτή, σε αυτή τη θητεία. Και είναι καλό, μια και η άλλη επιτροπή μου είναι η Επιτροπή Ενέργειας, είναι καλό να δει κανείς ότι υπάρχουν επικαλυπτόμενοι τομείς όσον αφορά τις αρμοδιότητες αυτών των επιτροπών όπως οι κλιματικές αλλαγές. Καλό είναι λοιπόν να συμμετέχω εδώ. Ευχαριστώ. Ik eh, heet Thijs Berman. Ik was journalist 20 jaar lang tot ευχαριστώ. Ήμουνα 20 χρόνια δημοσιογράφος. Πρωτού το 2004 ήρθα στο κοινοβούλιο. Ασχολήθηκα με την ε, γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μέχρι ότου κατέληξα εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Και πραγματικά το κυριότερο ενδιαφέρον μου είναι αυτό. Ενδιαφέρομαι ευρωπαϊκά αλλά και έξω ευρωπαϊκά για αυτή την ε, συνιστόσα για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι επικεφαλής και να δίνει σε όλους μια δυνατότητα. Και εδώ αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και το δυνατόν θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να είμαι χρήσιμος. Σας ευχαριστώ. Μάικλ Κάσμαν, μέλος ε, σε αυτή την Ευρωβουλή επί μια δεκαετία. Προηγούμενα στα ε, θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών και είχα ειδικευθεί στην, ε, στον ανοιχτό χαρακτήρα, στη διαφάνεια και στα δικαιώματα του ανθρώπου. Έχω τις εξής φιλοδοξίες. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε όλοι να είναι ίσοι σε αυτόν τον κόσμο. Η άλλη φιλοδοξία μου είναι οι πολιτικοί να μιλάνε λιγότερο και να πράττουν περισσότερα. Ευχαριστώ. Ο υπαριθμό 10 παρακαλώ. Uh, my name is uh, Πρόσιας Ντερόσα. Είμαι Ιρλανδός Ευρωβουλευτής ε, από το Εργατικό Κόμμα, μέλος ε, της Σοσιαλιστικής Ομάδας ε, και της Δημοκρατικής Σοσιαλιστικής Ομάδας εδώ. Είμαι κυριότερη επιτροπή μου. Είναι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων όπως τα τελευταία δέκα χρόνια. Και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος τομέας, ευρύτατος τομέας ε, ομοιοτήτων για αυτά τα θέματα που εσωτερικά τα αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, καθώς επίσης ομοιότητες σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πραγματικά πιστεύω ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί ώστε να διασφαλίσουμε ώστε οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη θα πρέπει να επιτευχθούν. Και ιδιαίτερα το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας που πρέπει και αυτό να επιτευχθεί. Είναι νομίζω ένας από τους πιο φιλόδοξους ε, τομείς ε, όσον αφορά τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια Πρόεδρε και συγχαρητήρια επίσης στους αντιπροέδρους. Είμαι ο Μιγελάν Μαρτίνερ Δέκα χρόνια ήμουν μέλο σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή και επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουν συντονιστή τη σοσιαλιστική ομάδα επίση. <clears throat> και ω αντιπρόεδρο τη Ευρωβουλή Είμαι ο συντονιστή των σοσιαλιστών αντιπροέδρων στο Προεδρείο τη Ευρωβουλής. Και μεταξύ άλλων πραγμάτων θα προσπαθήσω οπωσδήποτε όχι μόνο να συμμετάσχω στο δυνατόν ευρύτερα σε αυτή την Επιτροπή αλλά και να προασπίσω από το Προεδρείο της Ευρωβουλής όλες τις φιλοδοξίες και τους στόχους και τις ε, προσδοκίες ως στόχους αυτής της ε, εργασίας στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Είναι ένα όραμα που έχουμε για ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο που πρέπει να είναι η Ευρώπη να ασκεί έναν ε, ρόλο επιρροής όσον αφορά την ελευθερία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Hola, soy Enrique Guerrero Ενρίκε Γκερέρο είναι το όνομά μου, Ισπανό Ισπανός σοσιαλιστής, ε, νέο μέλος ε, στην Ευρωβουλή. Στο παρελθόν είχα αρμοδιότητες ε, στην ίδια την κυβέρνηση της Ισπανίας όσον αφορά τον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης και στον τομέα των σχέσεων μεταξύ της Βουλής και της κυβέρνησης του κυβερνητικού έργου. Και ο τελευταίος στόχος μου πριν από το να θελήσω να γίνω Ευρωβουλευτής ήταν ότι ήμουν αναπληρωτής επικεφαλής ε, του ε, γραφείου του ίδιου του Προέδρου της Ισπανική Κυβέρνηση, Πιστεύω ότι όπως αναφέρθηκε η συνεργασία και την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή μέσα σε μια συγκυρία κρίσης αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Αλλά έχουμε πιστεί ότι περισσότερο από οποιαδήποτε φορά ότι η ευημερία, η πρόοδος είναι αδιαχώρητα, είναι αγαθά που δεν μπορούν να διαρεθούν και πρέπει να ισχύουν για όλους, γιατί διαφορετικά δεν θα ισχύουν για κανένα. Πρέπει να ασκήσει την επιρροή της με κάθε τρόπο η Ευρώπη για να σημειωθούν πρόοδοι σε αυτούς τους τομείς. Ευχαριστώ. <clears throat> Το όνομά μου είναι Νόβερ Ρόιζερ. Προέρχομαι από τη Ρινανία Παλατινάτο στη Γερμανία. Είμαι νεοεκλεγέν μέλο. 18 χρόνια προηγούμενα ήμουν αναπληρωτής ε, ε, τοπικός ε, εκπρόσωπος Λάντρατ και στην συνεργασία για την ανάπτυξη με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μη κυβερνητικές ε, φορείς είχα συνεργαστεί. Μέχρι το 2014 ε, που κυρίως συμπίπτουν με τους στόχους της χιλιετίας 2015 στόχος μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας ετήσια να εξετάζεται και να μετράτε και χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Eh, Συγχαρητήρια Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, είμαι ο Ντάβιτ Σασόλη, έρχομαι από την Ρώμη, από την Ιταλία. Είμαι ο αρχηγός της αντιπροσωπείας του, Ευρωπαϊκού του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος και συμμετέχω στην ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είναι η πρώτη μου εντολή και πιστεύω ότι σε αυτήν την Επιτροπή έχουμε ένα στρατηγικό ρόλο να παίξουμε για την Ευρώπη. Να απαντήσουμε στην οικονομική κρίση δίνοντας ένα νέο νόημα στη συνεργασία και στην ανάπτυξη. Πιστεύω ότι εδώ παίζεται ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, δηλαδή του ότι η Ευρώπη θα, αποτελέσει, θα είναι κινητήρας ανάπτυξης και δικαιοσύνης. Euh, είμαι ο Πατρίς ε, Τυρολιά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είμαι ο Πατρίς Τυρολιά. Και είμαι εκπαιδευτικός. Δήμαρχος κιόλας. Στη Μαρή Γκαλόν, στη Γουαδελούπη. Σε ένα μικρό δήμο. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπώ την 8η εκλογική περιφέρεια των, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εγώ ήμουν περιφερειακός ε, σύμβουλος για θέματα οικονομικής συνεργασίας. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να προωθήσω τις ε, γαλλικές υπερπόντιες ε, περιοχές και πιο συγκεκριμένα τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα. Εγώ θέλω η Επιτροπή μας να ξεκινήσει μία πραγματική αναπτυξιακή πολιτική. Να δημιουργήσει ένα διεθνές αναπτυξιακό δίκαιο στο οποίο η Ευρώπη θα παίζει εξέχοντα ρόλο. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς και εκπροσωπώ την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πολλά χρόνια ήμουνα καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Επίση ήμουνα βουλευτή στην πατρίδα μου και τα τελευταία 25 χρόνια έχω εργαστεί με μη κυβερνητικέ οργανώσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ανάπτυξη σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Έχω λάβει τα μέρο ω χειρουργό σε όλου του πολέμου τη τελευταία 20 ετία και έχω δουλέψει σε πάρα πολλέ Αφρικανικέ χώρε, χώρε του Νοτιού Ειρηνικού, τη Ασία, τη Κεντρική Ασία, τη Καραϊβική, τη Λατινική Αμερική, ω θελοντή σε όλου του τομεί. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει εκτό από ηθική υποχρέωση απέναντι στον τρίτο κόσμο και δεν θα αναλύσω αυτή τη στιγμή του λόγου, και ουσιαστική υποχρέωση απέναντι στον ίδιο τη το λαό γιατί με την ανάπτυξη των χωρών των υποαναπτύρων χωρών των αναπτυσσομένων χωρών θα βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της μη ελεγχόμενης μετανάστευσης, των πανδημιών, των κλιματολογικών αλλαγών, τη ανάπλαση του περιβάλλοντος. Συνεπώς, ω Επιτροπή έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και θα είμαι στη διάθεση του Προεδρείου και τη Επιτροπή, για να ε, καταθέσω την εμπειρία που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Und auch meine Erfahrungen hier einbringen. Λέγομαι Τσαμπάν Ουρι, είμαι Ούγγρος. Από το 2004 είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, ε, είχα αναλάβει και μία εισήγηση, μία έκθεση. Έχω την πρόθεση να εργαστώ σοβαρά σε αυτήν την Επιτροπή για την επόμενη εκλογική θητεία. Ευχαριστώ. Σνίμπερ Γιάστραμ είναι το όνομά μου. Προέρχομαι από το Αμβούργο, μια μεγάλη πόλη στη Βόρεια Γερμανία. Για πρώτη φορά βρίσκομαι στην Ευρωβουλή. Πολιτική πείρα έχω από την Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία και ως ε, δεύτερη δημαρχίνα της ε, ελεύθερης και χανσεατικής πόλης ε, του Αμβούργου. Και έτσι μια σειρά αποστολών είχα κάνει υπό αυτή την ιδιότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το έργο το αναπτυξιακό και χαίρομαι να έχω συνεργασία μαζί σας σε αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι ο Κρήτανο Αρσένης, είμαι από την Ελλάδα νέο μέλος του Κοινοβουλίου στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Από τα 15 χρόνια μου είμαι στο περιβαλλοντικό κίνημα. Η ειδικότητά μου είναι η αηφόρος ανάπτυξη, αλλά και προφανώς και η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής του μοναδικού τόσο σημαντικού ζητήματος που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Οι σπουδές μου ήταν στη χωροταξία και στη διεθνή ανάπτυξη και πραγματικά θεωρώ ότι η Επιτροπή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί έχουμε αυτά τα πέντε χρόνια μπροστά λοιπόν, μα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και πραγματικά πώ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα οι αναπτυσσόμενε χώρε χωρί τη δικιά μα βοήθεια δεν έχουμε μέλλον σε ένα άνισο και άδικο κόσμο. Είναι πραγματικά η υποχρέωσή μα να, να διασφαλίσουμε ένα äh, αξιοπρεπή διαβίωση στου πολίτε όλου του πλανήτη, μια, την πρόσβαση σε, σε βασικά αγαθά, στο νερό, την αντιμετώπιση των ασθενειών, το ίσο δικαίωμα στη ζωή τελικά. Η πρόκληση που έχουμε πάει να δείξουμε είναι τεράστια και η ευκαιρία μοναδική. Και θα χαρώ να έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία να καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτόν τον äh, κόσμο. Ευχαριστώ uns liegt und ich hoffe, dass wir etwas verändern können. ευχαριστώ. Είμαι ένας από τους 7 βουλευτές της Σλοβενίας που εκπροσωπούνται στην Ευρωβουλή. Και γι' αυτό θα ήθελα να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία ώστε να πω και εγώ δύο λόγια στη γλώσσα μου, τα σλοβενικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για το ότι είμαι μέλος σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή. Γιατί όλη μου τη ζωή είχα αφοσιωθεί σε σχέση με τα αναπτυξιακά θέματα και ως υπουργό Εξωτερικών και πρέσβης της χώρας μου σε επισκέψεις σε διάφορες χώρες για αυτά τα θέματα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό λοιπόν. Πολύ σημαντικό να μην δημιουργήσουμε ένα οχυρό Ευρώπης, αλλά να δημιουργήσουμε γέφυρες από την Ευρώπη προς τις άλλες χώρες ώστε εκείνοι που επιθυμούν να προοδεύσουν να μπορούν να έρχονται στην Ευρώπη και να μην χρειάζεται μέσα σε σκαφίδια και πλοία και πλοιάρια να εγκαταλείπονται οι άνθρωποι και να προσπαθούν να περάσουν στην Ισπανία ή σε άλλες χώρες ε, αλλά η αναπτυξιακή πολιτική να δημιουργηθεί σε στερεές βάσεις για το μέλλον με τέτοια υποδείγματα ώστε όλοι ισότιμα να μπορούν να συμμετέχουν. Ευχαριστώ. Είμαι Βρετανό βουλευτή είναι Βρετανός βουλευτής, από τα East Midlands. Ο πιο γνωστός από την περιοχή μου ήταν ο ε, Ρομπέν των Δασών. Θα θυμάστε το σερίφι του Νότιχαμ που έπαιρνε από τους φτωχούς και μοίραζε στους πλούσιους. Συγγνώμη, από του πλούσιου και μοίραζε φτωχού. Είναι καλή αρχή αυτή για την Επιτροπή μα. Είμαι νέο στην Επιτροπή αυτή. Έκτη φορά είμαι Ευρωβουλευτή όμω. Είμαι πολύ παλιό Ευρωβουλευτή. Και είμαι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα τη αλλαγή του κλίματο. Πιστεύω ότι αυτά θα είναι χρήσιμα ως στοιχεία και για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και εγώ για την εκλογή σας ως Πρόεδρο. Από το 1994 μέχρι το 1999 ήμουν μέλο τη Επιτροπή ε, ε Ανάπτυξη. Λέγομαι Γκέρεν. Είμαι μέλο τη Ομάδα των Φιλελευθέρων. Έχω πέντε χρόνια θητεία υπουργό. Είμαι υπεύθυνο για το θέμα ανάπτυξης και ανθρωπιστική δράσης, περιβάλλον και για την άμυνα, αν σα φαίνεται κάπως περίεργο αυτό, είχα και αυτό το πόστο. Μετά έγινε πρόεδρος της ομάδας του για το Σαχέλ και της Δυτικής Αφρικής, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να συζητιώνται τα θέματα της περιοχής τη Δυτική Αφρικής. Όταν ήμουν υπουργό, είχα την ευκαιρία το Λουξεμβούργο να περάσει το 0,7% του ΑΕΠ για την ανθρωπιστική βοήθεια. Είχα βάλει στόχο το 1% του ΑΕΠ, το πλησιάζουμε, το 1%. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ζεμπού, ένας μεγάλος Αφρικανός σοφός που είπε «Δεν αναπτύσσει κανείς, αναπτύσσεται» αν καταλάβουμε αυτή τη φράση θα κάνουμε πολύ λιγότερα λάθη στην ανάλυση της κατάστασης των αναπτυσσόμενων χωρών. Επόμενος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας συγχαίρω. Λέγομαι Αρλέμ Ντεζίρ, είμαι Ευρωπαίος Σοσιαλιστής, εκλέγομαι στη Γαλλία. Είμαι αναπληρωτή στην Επιτροπή Ανάπτυξη. Στην κύρια Επιτροπή είναι το Διεθνέ Εμπόριο. Για μένα είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ εδώ και 10 χρόνια. 10 χρόνια είμαι βουλευτή η εμπορική μας πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική μας πώς συμφιλιώνονται, γιατί πρέπει να υπάρχει συνοχή και ακολουθία στη δράση της Ένωσης. Να μην από τη μια μεριά δωρητής, γενναιόδωρος και από την άλλη μεριά μέσω οικονομικών πολιτικών και ιδιαίτερα εμπορικών πολιτικών να ακολουθεί στενά εγωιστικά συμφέροντα. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς διεθνείς πρωταγωνιστής πρέπει να είμαστε πραγματικός εταίρος για τις χώρες του Νότου που σημαίνει πρέπει να συνδυάζονται οι εμπορικοί μας και οι μας στόχοι και πολιτικές. Και θα βοηθήσω σε αυτό. Ευχαριστώ. Όνομά μου είναι Γκάμπι Τσίμερ. Είμαι από τη Γερμανία. Είμαι Ευρωβουλευτήνα για το αριστερό κόμμα, τη Λίνκε στην Ευρωβουλή, δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία. Χαίρομαι να μπορώ να συνεχίσω το έργο στην Επιτροπή Ανάπτυξης με κέντρο βάρος στην καταπολέμηση της φτώχειας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φυσικά σε δέσμευση στην συνολική στρατηγική σφαιρικά για την ανάπτυξη και για τους στόχους της και για την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη συνεργασία στην ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ε, χαιρετώ για δεύτερη φορά. Λέγομαι Κατρίν Γκρέζ. Είμαι νεοεκλεγμένη πράσινη βουλευτής και μεγάλη μου τιμή πρέπει να πω ότι ε, εξελέγει η Εύα Ζολή πρόεδρος αυτής της Επιτροπής ε, αντιπροσωπεύοντας την ομάδα μου. Οι προτεραιότητες μου συνδέονται στα θέματα ανάπτυξης ε, και φοροδιαφυγής, ε, το πώς συνδέονται τα προβλήματα φοροδιαφυγής με την ανάπτυξη, το θέμα των αρρωσίμων γεών και γεωγραφικά ενδιαφέρομαι εγώ κυρίως ε, για τα θέματα ε, συντονισμού των πρασίνων παγκοσμίων, σε, κυρίως συνεργάζομαι με τη Λατινική Αμερική. Όνομα Κέλλα. Είμαι στην ομάδα των Πρασίνων, είμαι από τη Γερμανία και έτσι από το κόμμα των Πρασίνων στο Βραδενβούργο και ήμουν πρόεδρος των νέων Πρασίνων στην Ευρώπη και γι' αυτό εργαζόμουν μεταξύ, σε σχέση με τη, τους δεσμούς για την ανάπτυξη, σε σχέση με τη μετανάστευση. Και θέλω να τονίσω επίσης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ε, Καλό σα απόγευμα. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την Πρόεδρο για την εκλογή της. Είμαι ε, από την Ολλανδία. Ανήκω στην ομάδα της ΓΚΟΕ, της Ενωτικής Αριστεράς στην Ευρωβουλή. Έχω επανεκλεγεί και κατά την τελευταία θητεία είχα ασχοληθεί με θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων και γεωργία και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Χαίρομαι όμως ότι αυτή τη φορά μπορώ να εργαστώ και σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη. Σε αυτή την Επιτροπή νομίζω έχουμε πάρα πολλούς στόχους, πάρα πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, κλιματικές αλλαγές, αλλαγές κλιματική κρίση. Αν όλα αυτά όμως οδηγούν στο ότι κάποιες πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν ή δεν λαμβάνονται είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να εστιαστούμε σε αυτά. Και μπορούμε να συνεισφέρουμε νομίζω με αυτόν τον τρόπο για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα κατέβαλα προσπάθειες ε, για τα ναρκωτικά, για την καταπολέμηση των ε, ναρκωτικών όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες και τις επιπτώσεις των πολιτικών μας σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω θα μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσουμε αυτή την τάση για την λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τα ονόματα από εδώ, είμαι μακριά. Είμαι μέλος των Ολλανδών Πρασίνων Είχα εργαστεί στο τοπικό επίπεδο στην πολιτική στο Άμστερνταμ για τα τελευταία χρόνια και ήμουνα και δραστήρια για την αναπτυξιακή βοήθεια και όσον αφορά και τα θέματα της αφρικανικής πολιτικής. Είχα εμπλακεί σε σχέση με τη διαδικασία Κίμπερλι για τα ακατέργαστα διαμάντια και για τα θέματα εξορρυκτικής βιομηχανίας και θέματα εξόριξης ορυκτών μετάλλων καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Αγγόλα, Μοζαμβίκη ε, και των δίκαιων εκλογών και της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα προσέχω τα θέματα ανάπτυξης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και έτσι σε αυτή την Επιτροπή αυτό θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Ja, jag heter Isabella Lövin och ευχαριστώ από τη Σουηδία. Συμμετέχω λοιπόν στην ομάδα των Πρασίνων, λέγομαι Ισαμπέλα Λούβιν. 25 χρόνια εργάστηκα ως δημοσιογράφος στη Σουηδία. Βεβαίως έγραφα κυρίως για πολιτιστικά θέματα, αλλά τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με θέματα για το περιβάλλον. Και έγραψα και ένα βιβλίο σχετικά με την μείωση των ε, αλλιευτικών ε, πόρων. Ασχολήθηκα επίσης με τις σχέσεις ε, Σουηδίας και Ευρώπης. Ασχολήθηκα επίσης και με την Αφρική και τις ε, σχέσεις συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτησα επίσης και τις αλλιευτικές συμφωνίες που έχουν οι Αφρικανοί αλλιείς με την Ευρώπη και το τι επιπτώσεις έχουν για αυτούς αυτές οι συμφωνίες. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Επιτροπή Ανάπτυξης και ελπίζω να συνεισφέρω στις εργασίες της Επιτροπής μας. Με ενδιαφέρει το θέμα της αλλαγής του κλίματος και ελπίζω η Ευρώπη να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες μπορεί και να βοηθήσει σε επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέχασα κάποιον για τις συστάσεις των μελών, για τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, ξέχασα κανέναν. Όλοι εδώ, όλοι συστήθηκαν, ωραία. Θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την ποικιλομορφία των εμπειριών του καθενός στην Επιτροπή υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν βαθιές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και ελπίζω ότι όλοι μαζί θα επηρεάσουμε την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη, είναι ένα σημείο στα διάφορα. Λοιπόν, αν κάποιος έχει κάτι να πει και δεν μπορεί να περιμένει τη συνεδρίασή μας για αύριο, να το πει αμέσως. Αλλιώς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10.30 10 και μισή με 12.30 θα κρατήσει η συνεδρίαση. Προηγουμένως θα συνεδριάσουν όμως οι συντονιστές από τις 9 ως τις 10 και μισή. Παρακαλώ την δίκηση να αναφέρει σε ποια αίθουσα θα συναντηθούμε αύριο. PHS 1α2 σύμφωνοι. Ελπίζω λοιπόν να σας ε, συναντήσω όλους αύριο στις 10.30. Τελείωσε λοιπόν η πρώτη μας συνεδρίαση.